Um, παρακαλώ καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Γρήγορα, γρήγορα. Καθίστε λοιπόν παρακαλώ για να μην αργήσουμε και με την ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε μαζί σας και τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ξεκινάμε λοιπόν. Πολύ φασαρία κάνετε σήμερα. Τόμας, ευχαριστώ. Σημείο 1, αγαπητοί συνάδελφοι, έγκριση της μέσης διάταξης, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Σε ό,τι αφορά τις γλώσσες, υπάρχουν κάποιες γλώσσες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες δυστυχώς σήμερα και συγκεκριμένα τσεχικά, δανέζικα, εστονικά, φιλανδικά, κροατικά, λετονικά, λιθανικά, μαλτέζικα, σλοβενικά. Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Πείτε όποιοι δεν έχετε μαζί τις κάρτες σας. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία και πριν δώσω το λόγο και στον εισηγητή, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Λάβαμε μία δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από την Επίτροπο Γιούροβα. Την έχετε λάβει. Απλά εγώ θέλω να σας πω ότι Είμαστε όλοι εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχετε μια επιστολή από την Επιτροπή ΑΦΕΤ, γνωμοδότηση, όχι επίσημη όμως γνωμοδότηση, είναι μια απλή επιστολή που συνέταξε η Επιτροπή ΑΦΕΤ και δίνει τις απόψεις της. Δεν είναι γνωμοδότηση, αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη. συνάδελφοι κύριο που παρακολουθείτε το φάκελο, δεν είναι δηλαδή επίσημη γνωμοδότηση, είναι απόψη αυτής της Επιτροπής. Έχει διανεμηθεί σε εσά και αυτό το έγγραφο. Αυτό είναι ημερωτικά και τώρα θα παρακαλέσω τον εισηγητή. Αν θέλει το λόγο, εν συντομία, Γιάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ, αγαπητοί συνάδελφοι. Έξι χρόνια περίπου ε, συζητάμε το θέμα αυτό και βέβαια είχαμε και διαπραγματεύσει για μια γενική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε ό,τι αφορά την συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου. Υπάρχει επιτάπητος μια έκθεση που λίγο πολύ χρονολογείται από πέρυσι. Τώρα όμως και μετά από πολλές συζητήσεις συνοδεύεται και από συγκεκριμένες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο η ερμηνεία της συμφωνίας ε, να είναι ξεκάθαρη, να μην μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις παρερμηνείς. Θα προσαρτηθεί στη συμφωνία λοιπόν ε, το σχετικό κείμενο και θα δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα. Και θα είναι ε, διαθέσιμο στους ε, διαπραγματευτές. Διευκρινίζει τρία σημεία από τα οποία έχουμε επανειλημμένως τονίσει ό,τι αφορά την ελόγω συμφωνία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η συμφωνία αυτή και αυτό ήταν ε, εξ αρχή σαφέ, δεν αποτελεί νομική βάση για οποιαδήποτε μεταφορά συνοδεύει ε, τι υφιστάμενε νομικέ βάσει ε, στη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ή στι διμερεί συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτων μελών της Ένωσης. Άρα δημιουργεί ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όταν υπάρχουν ε, μεταφράσεις μεταβάσεις με βάση κάποια από αυτές τις ε, νομικές βάσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Δεν θεωρείται απόφαση καταλληλότητας ε, επηρεάζει ε, δεν έχει κάποια τέτοια ισχύ. Οι αρχέ προστασία των δεδομένων στα κράτη-μέλη πάντοτε έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το κατά πόσον τα πρότυπα συμμορφούνται με τα πρότυπα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χάρτη και φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι διατάξεις θα εφαρμοστούν και από την Αμερικανική πλευρά. Δεύτερο σημείο. Προβλέπεται ε, δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για τους πολίτες. Ε, πρέπει όλοι οι πολίτες να τα έχουν αυτά τα δικαιώματα. Αυτό είναι επιπρόσθετο σε πολλά άλλα δικαιώματα συλλογικών προσφυγών. Θα ισχύει πάντως και η συμφωνία αυτή στην προκειμένη περίπτωση ευρωπαϊκή πλευρά πίεσε την αμερικανική πλευρά να συμπεριλάβει και άτομα που είναι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι υπήκοοι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτό, δεν είναι δυνατόν. Ωστόσο, εγώ ερμηνεύω τα πράγματα ως εξής. Η συμφωνία αυτή από νομικής πλευράς λόγω της χάρτας και λόγω της συνθήκης θα είναι ε, έγκυρη και νομικά σε ισχύ παρότι δεν μπορεί, ή, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνει αυτή τη ρήτρα για τα δικαιώματα ε, των προσφυγών και αυτά το ένδικο μέσο που περιορίζεται προ το παρόν, επαναλαμβάνω, μόνο στου υπηκόου χωρών τη Ένωση. Αν στην Αμερικανική νομοθεσία υπάρξει οποιαδήποτε διάταξη η οποία περιορίζει τι διατάξει τη παρούσα συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει φυσικά ε, σε μια εφαρμογή τη συμφωνία αυτή. Και όπω προείπα ήδη, σημαίνει αυτό ότι η εν συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν έχει ισχύ. Ιδίως ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις στον νόμο περί ιδιωτικότητας ε, για τα αρχεία, ε, για το πρόγραμμα καταπολέμησης της και δημοκρατίας κτλ. Θα πρέπει λοιπόν η Αμερικανική πλευρά να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο αυτής της Διεθνούς Συμφωνίας, η οποία είναι και δεσμευτική. Με αυτές λοιπόν τις διευκρινήσεις και με την ασφάλεια δικαίου που έχουμε πλέον, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις ε, μεταφορές. Πολύ ε, βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση σε σχέση με σήμερα. Έχουμε πολλές ε, συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής. Εκεί οι διατάξεις για την προστασία δεδομένων είναι αρκετά μετριοπαθείς. Και εδώ έχουμε μεγάλη βελτίωση. Νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να δώσουμε την ε, σύμφωνη γνώμη μας, αυτή τη συμφωνία. Πρόεδρος, αυτή λοιπόν είναι η σύστασή σου. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε συζήτηση, αλλά υπάρχει ε, μια σύντομη παρέμβαση με την κυρία Ιντφέλτ επί της διαδικασίας. Κυρία Ιντφέλτ, θα ήθελα μια διευκρίνηση ό,τι αφορά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να είναι σαφές ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μιλάμε για τις εξαιρεσει από το Privacy Act, το νόμο περί ιδιωτικότητας. Λέει η Κομισιόν ότι με την λέει για την των εξαιρέσεων και θεωρεί ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή του άρθρου 91. Όπως απαιτείται και τα λοιπά, θεωρεί ότι το άρθρο 91 της Γενική Συμφωνίας αποτελεί μια ουσιαστική διάταξη της συμφωνίας που πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Συμφωνεί ο λοιπόν μαζί μου πως τούτο σημαίνει ότι εάν Εξαιρέσει έτσι οποίες συζητούμε δεν καταργηθούν, θα θεωρείτε ότι είπα δεν εφαρμόζουν την γενική αυτή συμφωνία. Σωστά ερμηνεύω τη δήλωση της Κομισιόν. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ωραία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, έρευνα, ανείχνευση και δίωξη ποινικών αδικημάτων. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Αν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν εφαρμόζουν τη συμφωνία συνολικά, οποιαδήποτε διάταξη. Δεν θα ξεκινήσουμε, λέει ο πρόεδρος, συζήτηση. Δεν θα ξεκινήσουμε συζήτηση. Η κυρία Ιντφελντ. Μα είναι βασικό. Είναι βασικό. Και χρειαζόμαστε διευκρίνηση. Γιατί τώρα ο λέει κάτι άλλο εάν αυτή η ερμηνεία της επιστολής είναι σωστή. Θέλω να ξέρω, Πρόεδρε, τι ψηφίζω. Ε, αυτή είναι η πληροφόρηση. Άρα, δημοκρατία, ψηφίζουμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Σας έδωσα το λόγο και ο εισηγητής απάντησε. Την δήλωση την πήραμε σήμερα, Πρόεδρε. Έλεος. Πρόεδρος. Έλα, Σόφη, τώρα. Πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Σύντομα παρακαλώ, σύντομα. Λοιπόν, να απαντήσω άλλη μια φορά. Αυτή η διευκρίνηση διευκρινίζει ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω η συμφωνία, ιδιαίτερα αυτό το σημείο. Αν δεν εφαρμόσουν οι ΗΠΑ αυτό το σημείο, τότε η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε από αυτού και είναι σωστό, αλλά και σημαντικό Επίσης επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμόσει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση αυτή την ε, συμφωνία και θέλουμε να υπάρξει αυτή η συμφωνία αν ε, συμμορφωθούν πλήρως με αυτήν και οι δύο συμβαλόμενοι. Ωραία λέει ο Πρόεδρος, τροπολογίες ένα και δύο ταυτόσιμες. Εντάξει είστε όλοι έτοιμοι. Άρχεται η ψηφοφορία από αυτόν. Βεβαίως και είστε έτοιμοι. Άρχεται. Έχασα την κάρτα μου. Καλά, λέει ο πρόεδρο. Καλά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ, γιατί είστε τόσο ε, και ανήσυχοι σήμερα. Η κυρία Γκόμες δεν έχει την κάρτα της, εντάξει το λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν την κάρτα τους. Η κυρία Γρισμπέκ και η Κορνέλια. Και δεν δουλεύει και το μηχάνημά σας. Μήπως μπορείτε να πάτε δίπλα. Παρακαλώ. Η κυρία Έρνστ θα χρησιμοποιήσει άλλη μηχανή ψηφοφορία και Γκόμες και Γκρισμπέκ δεν έχουν τι κάρτε του. Οκ, θα μα πούνε πώ θα ψηφίσουν. Εάν συμφωνείτε όλου. θα μα πούνε τι ψηφίζουν. Ε, παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, ο συγητής ε, θέλει να διευκρινίσω τι ψηφίζουμε. Αρχίζουμε με την παράγραφο 1. Έχουμε τις ε, ταυτόσιμες τροπολογίες 1 και 2 που είναι προτάσεις απόρριψης. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Ωραία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ, 40 κατά, 0 αποχές. Και τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 41 ψήφι υπέρ, 4 κατά, 6 αποχές. Συγχαίρουν τον εισηγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Έληξε η ώρα των ψηφοφοριών και περνάμε στα επόμενα θέμα της ημέρης διάταξης. Παρακαλώ να αποχωρήσετε αρκετά ησύχω για να περάσουμε στα επόμενα θέματα. Quietly, thank you. Colleagues, let's move to point four, which is the... Περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι σημαντικό. Καλά, να περιμένουμε ακόμη. Συντονισμός κάποιων ε, μέτρων ε, που, έχουν, ε, που ισχύουν λόγω μέσω νόμου κανονισμών ή διοικητικών ενεργειών και που αλλάζουν την κατάσταση όσον αφορά την, τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών. Ο μιλήτριά μας είναι η κυρία Μίλναρ. Θα παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ να κάνω μια σύντομη επισκόπηση της πρότασής μου. Είναι νέα προτάση που εγκρίθηκε τον Μάιο για να ενημερωθεί η νομοθεσία στις τεχνικές προσαρμογές και στις ανάγκες των καταναλωτών και δίνει περισσότερες δυνατότητες στις πλατφόρμες βίντεο για να καταπολεμήσουμε τα κηρύγματα μίσους και την διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου σε ανηλίκους αλλά δεν συμμετείχαμε στην προηγούμενη ε, οδηγία γιατί ήταν πριν να αρχίσει να ισχύει η συνθήκη του Λισαβόνα. και άρα ο χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είχε το ίδιο νομικό καθεστώ όπω οι συνθήκε. Η Επιτροπή μα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε μέτρο δικαστική συνεργασία για ποινικά θέματα και ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστεί ο ρατσισμό, η ξενοφοβία και οι ομιλίε μίσου. Όπω ξέρετε η γνωμοδότηση αυτή ήταν θύμα ε, σύγκρουσης αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή Κούλτ, την οποία χάσαμε αυτή τη μάχη. Όμως ε, πρέπει να εξαγάγουμε διδάγματα. Στο μέλλον πρέπει να επιδεικνύουμε περισσότερη συνέπεια και πάντα να υπερασπιζόμεθα τις αρμοδιότητές μας παρά τις πολιτικές πιέσεις συναδέλφων από άλλες επιτροπές. Τώρα, περιεχόμενο. Ω εισηγήτρια ασχολήθηκα με πέντε τομείς. Μια ισορροπημένη ε, προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το παράνομο περιεχόμενο, να διατηρήσουμε τις ε, εγγυήσεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, να είμαστε συνεπείς στην αντιμετώπιση του μίσους και της βίας, την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και τέλος και πολύ σημαντικό, ανεξάρτησία των ρυθμιστικών αρχών και σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Θα ασχοληθώ με αυτό το τελευταίο γιατί είμαι πεπισμένη ότι η ελευθερία του πλουραλισμού χρειάζεται τη βοήθειά μας. Επανειλημμένα ως Επιτροπή έχουμε καταδικάσει κράτη-μέλη και όχι μόνο για παραβιάσεις ανθρωπίνων συγγνώμη, θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το τομέα. Πρέπει τώρα όμως να κάνουμε κάτι παραπάνω, να δώσουμε δυνατότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δρά, για να αντιμετωπίζει παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ελπίζω να με στηρίξετε. Τέλος, ευχαριστώ τους Κιώδης να συνεργαστώ ε, προσβλέπω μαζί, μαζί τους για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ακουστεί η φωνή μας στην Επιτροπή Πολιτισμού. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιους σκιώδεις εδώ. Ο κύριος ε, Γκουάρου. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, σχετικά με την οδηγία των οπτικοακουστικών μέσων είναι πρόσδεκτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει ζητήσει την αναθεώρηση καθότι αλλάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά. Να πω επίσης ότι η οδηγία υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως και οι αρχές που είναι εγγεγραμμένες στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά λοιπόν στην προστασία των παιδιών, γενικότερα των ανηλίκων, αυτό είναι πρωταρχική σημασία για την ομάδα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να διατηρηθεί το ύψιστο επίπεδο προστασίας. Προστασία των παιδιών και ασφαλές περιβάλλον για την ανατροφή τους, αυτά είναι πρωταρχικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ε, το αναφέρει ξεκάθαρα εξάλλου το άρθρο 24. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει ως ε, Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για το ψήφισμα, για την προστασία των παιδιών ε, στον ψηφιακό κόσμο, έτσι ώστε να μην υπάρχει και ε, σεξουαλική τους εκμετάλλευση μέσω διαδικτύου. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι τα δικαιώματα των παιδιών ε, πρέπει να είναι προστατευμένα στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί επ' αυτού να υπάρχουν εξαιρέσεις. Και υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε σχετικά με το πρώην άρθρο 7 της οδηγίας ε, το οποίο διαγράφηκε αφαιρέθηκε από την τρέχουσα οδηγία. Ανέφερε αυτό και παραθέτω, οι πάροχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους ε, σταδιακά είναι προσπελάσιμες σε άτομα με ε, οπτικά και κινητικά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο για την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών και των ε, παροχών γενικότερα προς άτομα με προβλήματα όρασης. Μέχρι όμως να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά που ισχύουν, δηλαδή να ζητήσουμε από τα μέλη, να να προάγουν τη νοηματική, ε, την ε, ε, πλοήγηση, χειροκίνητη πλοήγηση, αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα νέο άρθρο της οδηγίας για τα μέσα ονημέρωσης. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις ε, προσπάθειές της και να τη διαβεβαιώσω ότι θα συνεργαστούμε μαζί της κατά το διάστημα που θα ακολουθήσει. είναι σκιώδης ηγητής ε, των σοσιαλδημοκρατών. Και εγώ συμφωνώ με τους προρελήσαντες ε, και εγώ καλωσορίζω αυτή την τροποποιημένη οδηγία. Η αγορά ε, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Και εγώ συγχαίρω την εισηγήτριά μας, την κυρία Μίλνερ, για την προσέγγιση της. Τα σημαντικότερα θέματα πράγματα εξετάζονται στο σχέδιο της γνωμοδότησής της. Όπως ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Ανεξαρτησία της έργα είναι καθοριστική σημασία σε αυτό για μας. Όσα έχει το πολιτικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτή η ανεξαρτησία είναι σημαντικότερη από ποτέ. Και από αυτού θα ήθελα να πω ότι εκτός ε, από το ότι πρέπει να διαδραματίζουμε καθοριστικό ρόλο, πρέπει πέρα από αυτό να κάνουμε και ό,τι μπορούμε για να μην υπάρχουν ιδιωτικές μόνο προσεγγίσεις. Δηλαδή ε, πρέπει οι ιδιωτικές αρχές να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους θέματα, αλλά όχι μόνο ε, να είναι αρμόδιος ο ιδιωτικός τομέας. Εγώ θεωρώ ότι η ε, αυτορύθμιση και η συνομοθετική δραστηριότητα είναι καθοριστική σημασία επί του θέματος. Αλλιώς είναι δυνατόν να υπάρξουν σημαντικές παραβάσεις του δικαιώματος ελευθερίας ε, θα μπορούσε να υπάρξει ε, εκμετάλλευση του περιεχομένου, κακή χρήση και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο και ο δισηγητής παρακαλώ. Ο Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ τον, την εισηγήτρια για την πολύ καλή πρόταση. Νομίζω ότι το σχέδιο της έκθεσης πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως με τη διαγραφή της λέξεως moral. Ε, έχουμε ε, θέματα όπως είναι αναλογικότητα και άλλα. Και ο χάρτης των δικαιωμάτων αναφέρει το άρθρο 15 πρέπει να γίνεται σεβαστό. Είναι πολύ σαφής αυτές οι διευκρινήσεις. Σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποια σημεία από τα οποίων έχουμε απορίες, για παράδειγμα. Ασφαλής νομοθεσία ή συνομοθεσία. Κομισιόν τα κράτη-μέλη. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Συμφωνώ. Πώς όμως. Νομίζω περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν για την την των σώμα των Ευρωπαίων ρυθμιστών. Κάποιες ε, άλλες τώρα ε, σκέψεις για την επάλυση της ηλικίας. Όποιο και αν είναι το σύστημα που θα ε, εφαρμοστεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε και τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχει μια δομή επιτήρηση παρακολούθησης Δηλαδή πάντοτε υπερισχύει το ότι δεν πρέπει να συλλέγονται παραπάνω προσωπικά δεδομένα πέραν των αναγκαίων. Σε ό,τι αφορά τη ρητορική μίσου στην τροπολογία 27. Σωστή η κατεύθυνση. Προστίθεται κατηγορίες στις λεγόμενες ευαίσθητες πληροφορίες, άλλα ευαίσθητα λεπτά θέματα όπως είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός κτλ. Ίσως να μην είναι πολύ ξεκάθαρο ακόμα το κείμενο, όμως στο τέλος γιατί λέει κάποια πράγματα για την ε, διάδοση ή διάθεση του ε, επιγραμμικού περιεχομένου. Πώς θα αποφασίζουμε, με ποια βάση θα περιορίζουμε τη διάθεση του οπτικού ακουστικού περιεχομένου. Πώς πρέπει να γίνει πιο σαφής ή πιο αυστηρή διατύπωση. για τον αποκλεισμό περιεχομένου. Και αυτό είναι ένα λεπτό θέμα. Έχει να κάνει με το πώς θα το οργανώσουμε. Και νομίζω ότι από διαδικαστικής πλευράς θα πρέπει να εμείνουμε στη θέση μας, δηλαδή να υπάρχει πάντοτε μία δικαστική μελέτη και ε, έγκριση Αυτέ τις παρατηρήσεις με γέννη όμως ε, είμαι ικανοποιημένο από την έκθεση και νομίζω ότι θα επηρεάσουμε και την ε, διαδικασία στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Και κυρίως πρέπει να μας πει το πώς θα προστατεύσουμε τους ανεξάρτητους ρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η Σκιώδης. Τώρα, ποιοι άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Ντόλτον, μην ανησυχείτε. Ήθελα να ακούσω πρώτα του Σκιώδη και τώρα εσεί είστε ο πρώτο ομιλητή. Αλλά είμαι Σκιώδη του ECR. Μα δεν το λέει εδώ αυτό. Με συγχωρείτε, δεν το λέει το χαρτί μου εδώ. Με συγχωρείτε, τώρα καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση, την εισηγήτρια και τα πολλά βήματα που κάνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης καλωσορίζω αυτά που γίνονται για να προστατεύσουμε τους ανηλίκου από λαβές περιεχόμενο και αυτού που μπορεί να θίγονται από τα κηρύγματα μίσου. Χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το επιβλαβέ περιεχόμενο ή οι παράνομες ε, ε, προτροπές προς ε, μίσο. Δηλαδή δεν πρέπει να το επεκτείνουμε πάρα πολύ πέρα από το φύλλο και το, τη θρησκεία, την εθνικότητα και το σεξουαλικό προσανατολισμό όσον αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογή. Δεν πρέπει να περιορίσουμε την περιορισμένη ευθύνη που είναι στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο για την ε, ελευθερία ε, έκφρασης και φυσικά πρέπει να προστατευτεί όπως ε, προτείνει και ο συγκεκριτής ανησυχώ για το ρόλο επιτήρηση που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Αυτέ είναι κρατικέ αρμοδιότητε. Και αυτό το έχει τονίσει και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Οι οπτικοακουστικέ υπηρεσίε βασίζονται στην αρχή της εδαφικότητα. Τα κράτη-μέλη ελέγχουν τι μπορεί να μεταδοθεί στην επικράτειά τους και τα δικαιώματα χορηγούνται σε εδαφική βάση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θίξουμε αυτές τις, ε, τις κρατικές ευθύνες και αρμοδιότητες. Συμφωνώ ότι πρέπει να αποσυρθούν κάποιοι όροι που είναι ανοιχτοί σε πολλές ερμηνείες αυτό τον όρο για την ε, ηθική ε, εκπαίδευση ε, και φυσικά δεν θα πρέπει να περιορίσουμε ιδιαίτερα την, την διάδοση του περιεχομένου. Και προσβλέπω στην δημιουργική συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους κοιόδης για να βρούμε τις σωστές λύσεις. Πρόεδρος. Δεν ενημερωθήκαμε ποιος εξέχων συνάδελφος του ECR είναι ο Σκιώδης. Τώρα ξέρουμε. Η κυρία Τσινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που έκανε σχετικά με αυτό το κείμενο το οποίο συζητάμε σήμερα. Και θέλω να ε, αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία επειδή εγώ είμαι και συμπρόεδρος από την Επιτροπή για τους ανήλικους, ε, για τους ανήλικες, για τα παιδιά, ότι πράγματι θα πρέπει όλοι οι ευρωπαϊκοί θυσμοί να εμπλέκονται στις διατάξεις και στους κανόνες που εγκρίνονται. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι σήμερα τα παιδιά, οι νέοι, οι έφηβοι που ζουν στην ψηφιακή εποχή, όλοι όλοι αυτοί ε, πολύ εύκολα μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο και να χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά προγράμματα. Αυτοί λοιπόν πρέπει να προστατευτούν. Και υπάρχουν ε, στατιστικά ε, στοιχεία από την Save the Children. Εκεί φαίνεται ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν κατανοούν τις ε, απειλές και τους κινδύνους που απεραίουν από το διαδίκτυο. Από την παιδοπορνογραφία μέχρι και άλλους πολύ σημαντικούς κινδύνους που έχουν σχέση με τη βία και την, τα κηρύγματα μίσους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά τη ε, Εγώ αυτό που ήθελα μόνο να επισημάνω είναι, όπως σας είπα, ότι πρέπει να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Λόρισον, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω την εισηγήτρια, επειδή εγώ έχω επαφές με δημοσιογράφους. Θέλω να σας πω ότι οι δημοσιογράφοι τα δέχτηκαν όλα αυτά με μεγάλη τους χαρά και θέλησαν και ο εμπορικός κόσμος να μπορεί κατά κάποιον τρόπο να ελέγχει το περιεχόμενο. Η θέση μας λοιπόν, ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός και χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες για την βία κατά των ε, παιδιών. Υπάρχει το περίπτωμα Euro Kids Online, ένας, ε, μια έρευνα που γίνεται και εκεί διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά είναι μόνα τους σε αυτή την εικονική πραγματικότητα είναι μόνο τους, ε, δεν επικοινούν με τους γονείς τους, οι γονείς ε, δεν ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά, ούτε και οι δάσκαλοι ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να ε, προστατευτούν ε, τα παιδιά χωρίς να υπάρχει κανένας ε, είδους εκπαιδευτική και γονεϊκή υποστήριξη. Αυτό είναι όμως το βασικότερο για να προστατεύσει κανείς τα παιδιά. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν εκείνοι που εργάζονται μαζί με τα παιδιά. Τώρα, για τη βία, οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε και αυτό φαίνεται από την έρευνα ότι το χειρότερο για τα παιδιά στα οπτικοακουστικά μέσα είναι οι ειδήσει, όπου τα παιδιά βλέπουν κάθε μέρα στην οθόνη τον πόλεμο, τη βία, ε, ας πούμε στη δική μου τη χώρα. Τα παιδιά 10 χρονών στο δημοτικό κλαίγοντας έβλεπαν τον Τραμπ να κερδίσει εκλογές και αυτό δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια γιατί για τα παιδιά ο Ντόναλτ Τραμπ είναι βία, ισούται με τη βία άρα δηλαδή βλέπουμε μια ατομική παρορμητική αντίδραση και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προστατεύονται παιδιά από αυτό το καθημερινό συναισθηματικό στρες. Εγώ σας το λέω πραγματικά εν είδη προειδοποίησης. Εμείς ε, εκπονούμε κάποιον κανονισμό, Καλό αυτό, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι τα πραγματικά προβλήματα βρίσκονται αλλού. Πανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που είπα στην αρχή. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, τα μεγαλύτερα αδέλφια, η ΜΚΟ, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και εδώ ε, καθοριστική σημασία είναι και η αυτορύθμιση. Εγώ υποστηρίζω ανεπιφύλακτα ότι θα πρέπει να στηρίζεται η αυτορύθμιση ε, και η επαγγελματική προσέγγιση και όχι ένας γραφειοκρατικός έλεγχος εκ των άνω. Λοιπόν, ε, απευθύνομαι στην εισηγήτρια το που ελέγχθη πράγματι είναι μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Συμφωνώ με όλα όσα ελέγχθησαν προηγουμένως. αυτή η έκθεση και το περιεχόμενο της έκθεσης ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που έχει και σχέση με την Επιτροπή Πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ε, θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα στους, σκιώδης, ε, στους συντονιστές, στους για να έχουμε μια πραγματικά καλή έκθεση. Και κατανοώ πλήρως αυτά που είπε εκ μέρους της Λίμπη ότι δεν θα είναι έτσι μια απλή έκθεση, ε, θα είναι μια έκθεση πολύ ισχυρή. Ξανατείνω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τα δικά σας Πρόεδρε και όλων των σκιωδών. Νομίζω ότι Είμαστε όλοι στο ίδιο μήκο κύματο. Έχουμε χρόνο για να ακουστεί η φωνή μα, για να συμπεριληφθεί και στην τελική έκθεση. Ε, βασίζομαι λοιπόν στη συνεργασία σα και χαίρομαι που όλοι ε, έχουμε τι ίδιε απόψει. Δεν θα είναι εύκολο να επιβάλλουμε την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Είχαμε μια ακρόαση στις Βρυξέλλες όπου η γνώμη των δύο εισηγητών της ΚΑΛΤ απήχαν πολύ από την δική μας θέση. Και όπως ε, είπατε και εσείς ε, κύριε Πάβελ, ε, είναι ζωτική σημασία στο θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν να με στηρίξετε. Δεν θα κατεβάσουμε τα χέρια. Δεν θα σταυρώσουμε τα χέρια. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Πρόεδρος, βεβαίως, βεβαίως. Ε, γνωρίζετε πολλά για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι η γνωμοδότηση θα είναι πολύ σωστή. Τροπολογίες μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 2 Δεκεμβρίου. Το τελευταίο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Ο εισηγητής ε, δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί. Αλλά η Άννα Γκόμες ε, ε, την ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε να τον αντικαταστήσει. Μια σύντομη εισαγωγή είναι τμήμα του πακέτου για τη μεταρρύθμιση του ασύλου. Και θέλουμε ε, αυτή, η, αυτό το γραφείο στήριξη του ασύλου να γίνει μια ε, απόλυτα ισότιμη με τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα μας πει κάτι για τις 582 τροπολογίες που έχουν πολιθεί και τι ε, περιεχόμενο έχουν. Δεν ξέρω τώρα πόσα σας έχει πει για όλες αυτές ο κύριος Νίλιο Μίλιο. Σας ευχαριστώ που τον ε, έχετε αντικαταστήσει και πέστε μου παρακαλώ πώς πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες. Κοιτάξτε, μου ζήτησε ο συνάδελφος ε, να πω τα εξής. Έξι από τις 84 ε, τροπολογίες ε, λάβαμε ε, σχετικά με αυτό τον κανονισμό για το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Ασύλου. Ε, με αυτή λοιπόν την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για τη συμβολή σας και από τις ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν καταλήγει στο ότι όλοι ε, υποστηρίζουν την γενική αυτή κατεύθυνση του σχεδίου της έκθεσης και μοιάζει να υπάρχει συμφωνία η ΕΑΖΟ να μετατραπεί σε έναν οργανισμό που θα αναλάβει ένα νέο ρόλο, δηλαδή να υποστηρίζει, να βοηθάει και να ελέγχει την εφαρμογή ε, της συμφωνίας CIS Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πάρα πολλές ε, δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τους οικονομικούς και τους ανθρώπινους πόρους. Είτε αυξάνοντας το προσωπικό αυτού του οργανισμού, είτε δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνεργαστεί με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες των Εθνών, έτσι ώστε να προσφέρεται τεχνική βοήθεια και άλλους βοήθεια στα κράτη-μέλη. Βεβαίως θα θέλαμε η ΑΖΟ να είναι πιο ευνοϊκή. Ο εισηγητής ε, θεωρεί ότι παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει, προστασίες και αυτά συμπεριλαμβάνονται στις τροπολογίες. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι η συνεργασία ανάμεσα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκών Συνόρων και Ακτοφυλακής. Η συνεργασία θα ενισχυθεί και οι φορείς αυτοί, οι οργανισμοί αυτοί θα είναι επίσης όρις. Είναι σημαντικό αυτοί οι οργανισμοί να κάνουν τις απαραίτητες αναλύσεις. Χαίρομαι που οι περισσότερες τροπολογίες είναι υπέρ του να προβλέπεται ένας καθοριστικός ρόλος για τον υποσυζήτηση φορέα έτσι ώστε να προσφέρεται βοήθεια στα κρατη για θέματα ασύλου, ε, να μην υπάρχει κλιμάκωση βίας και να μπορεί επίσης ο οργανισμός να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία του κοινού συστήματος χορήγησης ασύλου. Άρα δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο έλεγχος δεν είναι ικανοποιητικός αν δεν στηρίζεται από τον κατάλληλο μηχανισμό. Έχουν κατατεθεί πολλές απόψεις που συζητούνται. Ο Πίτερ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου οι σκιώδεις ηγητές θα καταλήξουν και θα είναι έτοιμοι η πρόταση έτσι ώστε να τεθεί σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ που αντικαταστά τον εισηγητή. Υπάρχουν κάποιοι σκιώδεις εδώ. Θα ήθελα κάποιο σε αυτόν τον λόγο. Κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Άννα για την έκθεση και να υπογραμμίσω ότι ο εισηγητή, ο Πέτερ Ντερμίλερ και οι υπόλοιποι σκιώδει έδειξαν ιδιαίτερη επικοδομητική στάση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αφενό είναι κρίσιμη σημασία αν θέλουμε να έχουμε μια, ε, ένα πλήρως ε, λειτουργούν ε, σύστημα παροχής ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί επίσης να εγγυηθεί ότι ένας θα μπορεί να έρθει στο ύψος των μελλοντικών προκλήσεων και να δείχνει με την απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να λάβουν την υποστήριξη. Αυτά που αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις ενώ ελπίζω μέχρι τα τέλη του χρόνου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Στο παρόν στάδιο θα ήθελα να επισημάνω τρία σημαντικά σημεία. Πρώτον, ο οργανισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στο να είναι στο δυνατόν πιο μεγάλη σύγκληση των αποφάσεων για την παροχή ασύλου, που σίγουρα είναι εθνική αρμοδιότητα και παραμένει. Ωστόσο, για να μην υπάρχει το λεγόμενο asylum shopping, δηλαδή να επιλέγει κανείς ε, τις πιο ευνοϊκές διατάξεις, θα πρέπει να έχουμε κοινέ διατάξεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν έχουμε πληροφορίε για τη χώρα προέλευση και σχετική κατάρτιση. ένα παράδειγμα. Δεύτερον, θα πρέπει ο οργανισμό να έχει τα μέσα ώστε να μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται βέβαια με ταχύ ρυθμού. μακριά από εθνικού εγωισμού. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μια δεξαμενή εμπειρογνωμόνων, αλλά και θα πρέπει να συνάπτονται συμφωνίε με οργανώσει που θα μπορούσαν Επίσης να παράσχουν βοήθεια. Τρίτον, χρειάζεται ένας ισχυρός μηχανισμός παρακολούθησης που θα αυξήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών Ασύλου και της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας θα αποτρέπει επίση μελλοντικέ κρίσει, εξασφαλίζοντα τη σωστή εφαρμογή του κοινού συστήματο παροχή ασύλου. Αυτό ο μηχανισμό θα αξιολογεί την δυνατότητα, την ετοιμότητα των εθνικών συστημάτων ασύλου και θα είναι ισχυρό. Που σημαίνει ότι θα μπορεί να επιβάλλει και κυρώσει στα κράτη-μέλη που ε, εκουσίω δεν εφαρμόζουν, δεν εφαρμόζουν το κοινό σύστημα. Δεν καταλαβαίνω πώ μπορούμε να δεχθούμε ένα κράτο μέλο να μην τηρεί τις δεσμεύσεις τους ό,τι αφορά το άσυλο. Αλλά παρόλα αυτά να εξακολουθεί να ε, απολαμβάνει τις ελεύθερες διακίνησεις μέσα στο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ που επόμενος ο μιλητής, ο κύριος ε, Άλλα Άχο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Γκόμες. Όπω υπόθηκε και σε προηγούμενε συζητήσει, η ομάδα μου ECR στηρίζει τη δημιουργία μια υπηρεσία ασύλου, εφόσον όμω θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στα κράτη-μέλη. Παράλληλα, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η ευθύνη τίμησης και προώθησης των αιτήσεων και επεξεργασία των αιτήσεων να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα κρατών μελών. Και δεν θέλουμε κοινή επεξεργασία των ε, αιτήσεων, ακόμη και αν το ζητήσει το κρατο μέλο. Παράλληλα, έχουμε επικρίσει για το ρόλο που προτείνουν πολλέ τροπολογίες για τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στι συμβαστικέ. Η μετανάστευση είναι πολιτικό θέμα και η πολιτική ιδιαιτερότητα των μη καπαόμικρων είναι ιδιαίτερα συζητήσιμη. Θα προτιμούσαμε να απαλληφθούν οι αναφορές στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου στην μετεγκατάσταση των προσφύγων και των τον άσυλο. Δεν θεωρούμε ότι η μετακατάσταση είναι λύση για το μεταναστευτικό. Στόχος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και τη αντίστοιχη υπηρεσία που θα είναι ένα μέσο αυτής της πολιτικής θα έπρεπε να είναι να αποφευθεί η επιλογή χώρας ε, υποβολής ε, αιτήσεων και ε, να μην διευκολυνθεί το σύστημα ΣΥΡΟΥ να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μετανάστευσης. Κατά τη γνώμη μας, πολλές συμβαστικές τροπολογίες δεν βελτιώνουν την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν όχι, Άννα, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω τον κύριο Κόλλιο που είπε ότι μια χώρα η οποία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το σύστημα χορήγης ασύλου θα πρέπει να ε, αποκλείεται, να εκδιώκεται από τη Συμφωνία Σέγγεν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το πω και στον Πίτερ, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Να αναφέρω μια άποψη που είναι του Πίτερ, Δηλαδή είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την επικάλυψη εργασιών ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνόρων και Ακτοφυλακής με τον νέο Οργανισμό ε, Χορηγής Ασύλου να μην υπάρχει επικάλυψη εργασιών. Ο ρόλος ε, αυτού του δεύτερου οργανισμού, του υποσύσταση, είναι να διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων και των νόμων. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα μπορεί αυτός ο νέος οργανισμός να λέει στα κράτη-μέλη, ε, στην περίπτωση που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις, ότι οφείλουν να τις τηρούν. Και δεν μιλάω τόσο για το θέμα της επεξεργασίας των ετοιμάτων ε, χωρίς ασύλο, αλλά υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάρη η Ελλάδα. Η Ελλάδα προφανώς ε, βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ως γνωρίζουμε, η Ελλάδα δεν είχε οργανισμό για να ασχοληθεί με όλα αυτά, αλλά είναι ανησυχητικέ κάποιες περιπτώσεις όπου η βοήθεια η τεχνική αρρωγή αν θέλετε, η βοήθεια ε, του οργανισμού θα μπορούσε να είναι καθοριστική σημασία. Ήμουνα πρόσφατα στην Ελλάδα με τους υπαλλήλους της ΕΑΖΟ και εμείς βοηθήσαμε τις ελληνικές αρχές ε, στην ε, μετεγκατάσταση, επεξεργασία αιτήσεων για μετεγκατάσταση προσφύγων. Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και ο ρόλος του ΕΑΖΟ θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερο προσωπικό, όπως το έχουν υποσχεθεί στους Έλληνες. Αλλά τι να το κάνουν το προσωπικό. Λένε οι Έλληνες το ισχυρίζεται τουλάχιστον όταν ο ρόλος του Άζο έτσι κι είναι περιορισμένος. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Είναι κάτι που πράγματι πρέπει να προβάλλεται. Και εξάλλου είναι σημαντικό και όταν πρόκειται και για τις προϋποθέσεις κατάσταση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο ελέγχθη. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. 8 Δεκεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ την Άννα, τους ε, Σκιώδης και συνάδελφοι. Τελειώσαμε. Δεν ξέρω στα διάφορα αν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Επόμενη συνάντηση είναι στις 29 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.